Chers collègues, la séance est ouverte. Je Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θέλω να καλωσορίσουμε και πάλι την ε, Μεριάντα. Το καλό των εκλογών είναι ότι είστε και πάλι μαζί μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε απόψε. Να σας πω ότι δεδομένων των δεσμεύσεων ε, του συναδέλφου Ολμπρίχτ θα ψηφίσουμε το 12 μετά το 8. Αν ε, δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρώ πως ε, συμφωνείτε με αυτή την ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 21ης Νοεμβρίου βρίσκονται στο φάκελο της ε, συνεδρίασης. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε πως αυτές οι αποφάσεις γκρίνονται. Και τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω δύο σημαντικά νέα ε, η ομάδα των σοσιαλιστών όρισε τον κύριο Βλαδιμίρ Μάνκα ως εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού για το 2020 και το ΕΛΚΑ την Μόνικα Χολμάγερ ως γενική εισηγήτρια για το τμήμα 3. Εάν λοιπόν ε, θέλετε να κάνετε στοιχήματα, να βάλετε στοιχήματα για τις πιθανότητες εκλογής του κυρίου Μάγκα και της κυρίας Χολμάγερ, νομίζω πως είναι μια καλή τοποθέτηση. Χαιρετίζουμε λοιπόν εκ των προτέρων την επανεκλογή τους. Λάβατε το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίας της 21ης Νοεμβρίου. δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρώ ότι αυτά τα πρακτικά εγκρίνονται. Απόψε έχουμε μια ιδιαίτερα φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο που θα μας απασχολήσει για κανένα μισάωρο είναι για να σας πω με ποια ανακούφιση πριν από μία μόλις εβδομάδα, ε, στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου που έπρεπε να αποφασίσει η νέα εκδοχή του σχεδίου προπολογισμού 2019, διότι η συνδιαλλαγή είχε αποτύχει, ε, αυτή η νέα πρόταση υποβλήθηκε στην Επιτροπή μας από τον Επίτροπο Οτίνγκερ στις 3 Δεκεμβρίου. Ε, συνεδριάσαμε με το Συμβούλιο σε τριμερή το 4 και αυτός ο τριμερής που τελείωσε αργά το βράδυ λίγο πριν ε, τα μεσάνυχτα, όχι και τόσο αργά, μας επέτρεψε μια προσωρινή συμφωνία που υποβλήθηκε στους συντονιστές μας στις 5 Δεκεμβρίου. Υπευλήθη στην Κορεπέρ στις 7 Δεκεμβρίου η οποία ο Κορεπέρ με τη σειρά της ε, εξέδωσε θετική γνώμη πριν να περάσει στη ψηφοφορία για τις δημοσιονομικές τροπολογίες για τη θέση του Συμβουλίου στη συναποψινή ψηφοφορία. Θα πρότεινα να ακούσουμε τον γενικό μας συζητητή Ντανιέλε Βιώτη που ε, ολοκλήρωσε μια φανταστική δουλειά με τους συναδέλφους Ρούμπεκ και Γκάγερ, με τους Κιώδης, με τους πολιτικούς συμβούλους, με όλα τα μέλη της συνδιαλλαγής, διότι κατά βάθος ήταν ε, πολύ ε, θετικό το ότι αυτή η συνδιαλλαγή ολοκληρώθηκε και μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στο, θετικά στον τριμερή της 5ης Δεκεμβρίου. Έχετε το λόγο κύριε Γενική Εισηγητά. Presidente, ringrazio, <clears throat> ringrazio le colleghe e colleghi presenti. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι σήμερα παρόντες και με βάση τόσο είπατε στο τέλος να πω και εγώ ότι αυτή δεν είναι επιτυχία του Γενικού Εισηγητή ούτε μόνο των ε, εισηγητών ε, των άλλων κατηγοριών και των οργανισμών ούτε των σκιωδών μόνο. Πιστεύω πως αυτή η επιτυχία που εντός λίγο θα σας την περιγράψω ε, είναι ένα επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ε, επιτυχία αυτής της Επιτροπής ε, των Ευρωβουλευτών που έδωσαν εντολή πολύ ισχυρή και ξεκάθαρη σε δύο διαφορετικές ε, ευκαιρίες, τρεις μάλλον, Μάρτιο, Ιούλιο και έπειτα με την ψηφοφορία της ανάγνωσης του Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό. Έλεγα λοιπόν ότι αμέσως έδωσα μια γνώμη για τη συμφωνία που την όρισα ως επιτυχία γιατί το αίτημα που υπέβαλε το Ευρωκοινοβούλιο επανελειμμένα προς ε, τον Γενικό Εισηγητή και προς την διαπραγματευτική ομάδα ήταν να έχουμε μία, ένα σημαντικό πολύ σημαντικό αντιστάθμισμα σε σχέση με αυτό που εμείς ε, θεωρήσαμε ως ε, αποτυχία του Συμβουλίου απέναντι στο θέμα του μέσου για τους προ... Σύριους πρόσφυγες στην Τουρκία. Δηλαδή, ένα δις από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού... της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτό το μέσο, χωρίς να ζητήσει την γνώμη του άλλου σκέλους ε, που είναι αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή του Κοινοβουλίου. Το αίτημα ε, που υποβάλλατε στην ε, διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ήταν ότι για το ένα δις για αυτό το μέσο να έχουμε ένα δις φρέσκο χρήμα για τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, δηλαδή για τις κύριες γραμμές για τις οποίες στηρίζει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το αποτέλεσμα το πετύχαμε, πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν γιατί με βάση τη συμφωνία που έγινε γίνεται μια αύξηση των γραμμών των δαπανών του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ε, για 45,3 ε, ε, εκατομμύρια. Βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία, υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος και αυτό δεν μπορούμε παρά να το πούμε μεταξύ μας, διότι υπάρχει, πώς να το πω, και το λέω με μεγάλη ταπεινότητα, υπάρχει και μια ήττα δική μας. Διότι όταν τον Οκτώβριο ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιμένει, η Επιτροπή θέλησε να εισάγει στην ε, συζήτηση και στην πρόταση της συνδιαλλαγής ε, την ενεργοποίηση του άρθρου 15 3 είναι αυτό το περίφημο άρθρο επί το οποίο έχουμε πια πει ότι ήταν να υποθεί, έχουμε πει άπειρα λόγια αυτές τις εβδομάδες, είχαμε την ε, δύναμη να υπερασπιστούμε την ενεργοποίηση εκείνου του άρθρου. Δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί για να ζητήσουμε αυτό το άρθρο να ενεργοποιηθεί και να υπάρξει για πρώτη φορά η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε χρήματα που δεν έχουν δαπανηθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και να τα κατευθύνουμε στις δαπάνες για την έρευνα ε, μας πιαστήκαμε προτίμαστε εμείς και το Συμβούλιο και ε, στην προετοιμασία αφιερωθήκαμε στο να καταφέρουμε τουλάχιστον αυτό εγώ καταλαβαίνω από το τελικό αποτέλεσμα του προπολογισμού. Όσο γίνεται περισσότερες επενδύσεις για τους πολίτες μας, αντί να σταματήσουμε και να επιμείνουμε για μια αρχή. Πιστεύω πως κάναμε σωστά, Πρόεδρε, όταν μαζί ως αντιπροσωπεία στην πρώτη συνδιαλλαγή αποφασίσαμε να σταματήσουμε την διαπραγμάτευση. Και αυτό γιατί δεχτήκαμε επίθεση από πλευρά του Συμβουλίου. Υπήρξε μια απόπειρα να μας εκμηδενήσουν και δείξαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα και αν δεν κατάφερε να, να επιτύχει όλα όσα επιθυμούσε από την άποψη των αρχών, τουλάχιστον κατάφερε να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα όσον αφορά την οικονομική συμβολή προς το μέλλον Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω άλλο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και ήσασταν πολύ ευγενικοί, με ανεχτήκατε και με στηρίξατε σε κάθε φάση. Έχετε δει όλα τα έγγραφα, τα έχετε, ξέρετε ποιε ήταν οι κινήσει και ξέρετε και ποιε είναι οι αυξήσει που πετύχαμε, ποιε είναι οι δεσμεύσει που θα έχουμε για την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν νομίζω πως αυτή είναι η γνώμη μου, ότι δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να υπερψηφίζουμε και αυτό ζητώ και από την ε, Επιτροπή μας. Φυσικά με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και τις πολιτικές απόψεις των ε, πολιτικών ομάδων, όμως νομίζω πώς μπορούμε να αρχίσουμε να υπερψηφίζουμε αυτή την συμφωνία για τον προπολογισμό του επόμενου έτους με ψηλά το κεφάλι και εφόσον προσπαθήσαμε να κάνουμε το maximum για να υπερασπιστούμε τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου και να μπορούμε επίσης να σταθούμε ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών με περισσότερους πόρους, πολύ περισσότερους πόρους από ό,τι αρχικά αναμέναμε στην αρχή της φάσης της συνδιαλλαγής. Αν θέλετε μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικό, αλλά πιστεύω πως ήδη είμαστε αρκετά κουρασμένοι να μιλάμε, έχουμε βαρεθεί να μιλάμε για αυτά τα νούμερα, τα έχουμε διαβάσει ξανά και ξανά και ε, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci, Ευχαριστώ, κύριε Γενική Εισηγητά. Επομένως, ακούστηκε η θέση μας και καταφέραμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτελέσμα. Και αυτό το καταφέραμε γιατί η διαπραγματευτική ομάδα ήταν ισχυρή και ήταν ισχυρή γιατί ήταν ε, ενωμένη. Ο Πόλο Ριουμπίχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τον γενικό μας ε, εισηγητή, τον κύριο Βιώτη. Ήταν πραγματικά επίμονος, υπέβαλε πολλές προτάσεις και ε, τελικά καταλήξαμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αρτούη, που έμεινε μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και που επίσης συνέβαλε στο να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούσαμε να αποδεχθούμε και να υπερψηφίσουμε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Γκάιερ, του οποίου επίση η συνεισφορά ήταν πολύ ε, σημαντικά. στην κεφαλίδα 5 καταφέραμε 2,9% στις ε, πιστώσεις καταφέραμε η αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να παραμείνει αμετάβλητη, ο προπολογισμό της δηλαδή, και έτσι το Συμβούλιο επίσης προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και υπήρξε και μια θεωρητική περικοπή ε, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ήταν μια συμβολική αν θέλετε περικοπή την οποία μπορέσαμε να ε, αποδεχθούμε. Λάβαμε και τις πέντε επιπλέον θέσεις για ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά μισό εκατομμύριο επίσης αυξήθηκαν οι πιστώσεις για τα πληροφορικά συστήματα και επίσης για την Ευρωπαϊκή Περισσορία Εξωτερική Δράση ε, πήραμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τι στρατηγικέ δράσει επικοινωνία. Επίσης, ε, μα υπόθηκε βεβαίω ότι θα γίνουν περικοπές 4,2 εκατομμυρίων ευρώ για ε, πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν, 750.000 ευρώ περικοπές είχαμε για την κτηριακή πολιτική. Ήταν αλλαγές τις οποίες καταφέραμε να αποδεχτούμε γιατί ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε προϋπολογισμό για το 2019. Ξέρετε ότι οι χρονιές στι οποίες γίνονται εκλογές είναι πολύ κρίσιμες, είναι δύσκολες. Γι' αυτό και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι καταλήξαμε εν πάση περιπτώσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε και επιδείξαμε ε, μια ενωμένη στάση εδώ ε, και το ότι όλες οι προσπάθειές μας κατευθύνονταν προς τον ίδιο στόχο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Merci σας ευχαριστούμε διότι βρήκατε τις σωστές λέξεις, τις ακριβείς λέξεις για να πείσετε την Αυστριακή Προεδρία, κύριε Ρούιμπιχ. Ο Γιάννης Γκάγερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, με όλους τους ε, ε συναδέλφους. Μια διαδικασία που ε, ε, είναι παράδοση άλλωστε σε εμάς είναι πάντοτε πολύ σημαντικό να μπορεί μια διαπραγματευτική ομάδα να προσέρχεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με ενωμένη φωνή. Από αυτή την άποψη λοιπόν θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν συμπεριλαμβανομένων όλης της ομάδας, των συναδέλφων, των βοηθών, των πολιτικών ομάδων. Με, τις, με τους οργανισμούς η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν κάπως ενδιαφέρουσα γιατί συνέβη κάτι σχετικά συνήθιστο στις διαπραγματεύσεις. Η αρχική θέση του Κοινοβουλίου ε, ήταν πολύ πιο κοντά σε εκείνη του Συμβουλίου παρά σε εκείνη της Κομισιόν. Να το πω διαφορετικά, ε, είχαμε μια συνεννόηση, να το πω έτσι, με, τις, ε, με εκπροσώπους του Συμβουλίου. Η δε Κομισιόν ήταν κάπως επιφυλακτική. Αλλά ε, όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται προς ε, τους οργανισμούς, είχαμε την κοινή θέση με το Συμβούλιο ότι αφού διευρύνονται οι αρμοδιότητε του, θα πρέπει αυτό να το εκδοπρίζεται και στους πόρους που κατευθύνονται σε αυτούς. Η Κομισιόν δεν ήταν ότι διαφωνούσε, αλλά ήταν κάπως πιο επιφυλακτική. Ε, για τους οργανισμούς υπήρξε και μια, ένα παζάρεμα, να το πω έτσι, χωρίς όμως να καταλήξει ε, σε μια γενικότερη συνολική μάλλον ε, αύξηση των κονδυλίων. Καταλήξαμε λοιπόν στο να υπάρξουν κάποιες περικοπές μόνο αν και εφόσον στην πορεία του 2019 φανεί ότι δεν χρειαστούν ή εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί και σχετική νομική βάση. Εμείς είπαμε ότι ε, άπαξ και δημιουργηθεί η νομική βάση και άπαξ και παρουσιαστούν τέτοιες ανάγκες ή τέτοιες δυνατότητες περικοπών μπορούμε μετά την ε, συγκρότηση σε σώμα του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε τέτοιες περικοπές. ήταν το γενικό σημείο που κρατάμε είναι ότι οι περισσότερες προτεραιότητες μας αναγνωρίστηκαν. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά ε, δεν καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό με το οποίο διαφωνούσαμε, να διαγραφεί δηλαδή αυτός ο στόχος περί 5% περικοπών του προσωπικού. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο σε όσους από τους σκιώδεις εισηγητές είναι παρόντες και θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Τάραντ για παράδειγμα και είναι παρόν και ενδεχομένως θέλει το λόγο να μοιραστεί μαζί μας τις εκτιμήσεις του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι πέρασα όλο το Σαββατοκύριακο εξετάζοντας τις επιλογές μου, διαβουλεύτηκα με τους δημοκράτες των χριστιανών δημοκρατών, τους δημοκράτες των σοσιαλιστών δημοκρατών, τους δημοκράτες των φιλελεύθερων ακόμα και αποφάσισα να μην χρησιμοποιήσω το πυρηνικό μου όπλο και να μην υποβάλω τροπολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί αλλιώς θα μας υποχρεώνατε να ψηφίσουμε εναντίον του άρθρου 15.3. Θα το θέταμε εν κινδύνο Α. Σας ευχαριστώ λοιπόν που συμβάλατε για να αποφύγουμε τη διάσπαση της ομάδας μας και χαιρετίζω την σοφροσύνη σας. Κυρία Μυριάντα, ο προϋπολογισμός σας ταιριάζει. Κοιτάξτε, με κανένα προϋπολογισμό δεν θα είναι κανείς ευχαριστημένος 100% αλλά θέλω να, συγχω... να συγχαρώ όλους όσοι έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια συγκεκριμένη γραμμή για την άμυνα. Η μεγαλύτερη υπαρξιακή αλλαγή, ε, απειλή είναι η κλιματική αλλαγή ούτω ή άλλως και χαίρομαι για όσα συμπεριλαμβάνονται προ αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να συγχαρώ ε, όλους όσοι δούλεψαν. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ. Επομένω, λέει ο πρόεδρο, τις επόμενες ημέρες, πριν τα Χριστούγεννα, είστε έτοιμοι να δουλέψετε πάνω σε μια νέα συνδιαλλαγή θα μπορούσα να ε, πιστώ, ίσως καταφέρετε να με πείσετε, Ε, οι τροπολογίες που έχετε υποβάλει είναι πληθωρικές. Και αν έστω και μία ψηφιστή, θα κάνει το, το, συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στο τριμερή διάλογο να καταρρεύσει. Ε, χαριτολογώντας το λέω. Η κυρία Γκάρτια Θαμπάλ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι πολύ βεβαρημένη η ημερήσια διάταξη, θέλω και εγώ να είμαι σύντομη και γι' αυτό θα συγχαρώ όσους εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια καλή συμφωνία παρά τα προβλήματα που είχαμε και ενδεχομένως είναι και η καλύτερη συμφωνία ε, σε όλη την ιστορία των προϋπολογισμών των ε, τελευταίων ετών. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε όλους όσοι ε, δούλεψαν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα η θητεία μας θα ολοκληρωθεί με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Είχαμε ξεκινήσει με αποτυχία στη συνδιαλλαγή το 2014 και ολοκληρώνουμε τη θητεία με άλλη μια αποτυχία στη συνδιαλλαγή, αλλά επιτυχία στον τριμερή διάλογο. Και αυτό είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να συγχαρώ όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή. Συγχαίρω τη γραμματεία την ομάδα της Γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών που έκανε εξαιρετική εξαιρετική δουλειά και θα ήθελα όλοι να τους χειροκροτήσουμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της γραμματείας λοιπόν. Bon, il est... Είναι 8 η ώρα και θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μετά το Brexit και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυρία Κάρτια Θαμπάλ. Υιοθετώντας την απλουστευμένη διαδικασία για τη νομοθετική διαβούλευση με το Συμβούλιο. Θα πάρει το λόγο για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι από τις ψηφοφορίες που ποτέ δεν θα ήθελα να είχαμε, γιατί πρέπει να προσαρμοστεί το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Ωστόσο, όπως πάντοτε, οφείλουμε να ε, ε, προνοήσουμε και η γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με την τροποποίηση της συμμετοχής των κρατών μελών στο ε, κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εν ώψη της μελλοντικής πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ε, για το ότι όπως πολλές φορές έχει υποθεί στους, εντός αυτής της Επιτροπής ζητούμε από τα κράτη-μέλη το εξή. Άπαξ και αποχωρεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το κεφάλαιο που θα διαφύγει να αντικατασταθεί από νέο κεφάλαιο από τα υφιστάμενα κράτη-μέλη για να μην μειωθεί η επενδυτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει αυτή την απόφαση, επομένως αν όλα γίνουν έτσι όπως έχουν προβλεφθεί, κάποια στιγμή στο μέλλον θα έχουμε αυτή την πρόταση συμπλήρωσης του κεφαλαίου του κεφαλαιακού αποθέματος της τράπεζας, της κεφαλαιακής επάρκειας μάλλον, την οποία θα, το κομμάτι αυτό θα χάσουμε λόγω της απαχώρησης του Εμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος. Επομένως μας καλείται να εκφέρουμε θετική γνώμη στην πρόταση αυτή, όταν θα μας έρθει. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Ποιος θα ήθελε να εκφράσει την απόψή του για το θέμα αυτό. Ο κύριος Βουάρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη συνεδρίαση, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες της πρότασης. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ούτως ή άλλως θα ισχύσουν εφόσον και αν τελικά αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία ψηφοφορίας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να μην φανεί το όνομά μου ως ε, κάτι που εγώ θα στηρίζω. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απέχω. Το σημειώνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Πράγματι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να εκφράσει γνώμη παραμονής την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 29 Μαρτίου και αυτό είναι δυνατό και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Επομένως αυτό σας καθησυχάζει κύριε Σουάρτς. Είναι η θέση του δικαστηρίου. Ε, μας την ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο. Καλώς. Άρα μπορώ εγώ να θεωρήσω ότι ο κύριος Βουάρτ δεν θα συμμετάσχει, θα απέχει. Αλλά δεν είναι ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρήσω ότι η γνωμοδότηση μας προτείνει η κυρία Γκαρτία Σαμπάλ εγκρίνεται από την Επιτροπή Προϋπολισμών. Κύριε Τάραντι, είστε εντάξει? Κανένα σχόλιο. Είναι πολύ καλή πρόταση. Θέλω να δείξω τη στήριξή μου. Δεν έχω τίποτα να πω. Αν δεν ε, μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο και ούτως ή άλλως χάνουμε και απέχει δηλαδή. Καλώς, άρα θεωρώ ότι η Επιτροπή μας ακολουθεί τον εισηγητή. Τώρα λοιπόν θα αποφανθούμε για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού που έχουν να κάνουν με τη θέση του Συμβουλίου έτσι όπως εγκρίθηκαν στη Κορεπέρ της 7ης Δεκεμβρίου. Μιλούμε για το προσωρινό, ε, ε, την προσωρινή συμφωνία. Θέλουμε το σχέδιο προπολογισμού να εγκριθεί αυτή τη βδομάδα και πρέπει για να γίνει αυτό να καταψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες γιατί αν ψηφιστεί έστω και μία τροπολογία η συμφωνία θα καταπέσει. Πάρα πολλέ ε, τροπολογίε έχουν υποβληθεί και έχουν βρει το δρόμο τους για την Ολομέλεια και όλες αυτές από μία πολιτική ομάδα. 11 τροπολογίες κατατέθηκαν στη γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών από την ίδια πολιτική ομάδα. Ένας κατάλογος ψηφοφορίας με μορφή αρχείου Excel σας έχει διανεμηθεί. Προτείνω να ψηφίσουμε σε μπλοκ όλες τις τροπολογίες και η ένδειξη του εισηγητή είναι να τις καταψηφίσουμε στο σύνολό τους. Γιατί αν έστω και μία τροπολογία εγκριθεί, η συμφωνία θα καταπέσει. Άρα, να έχουμε 10 λεπτά έγκαιρη ενημέρωση για το σχέδιο πτήσης και το σχέδιο ψηφοφοριών. Για την ψηφοφορία λοιπόν on block, στο σύνολο, σε block, δεν βλέπετε κάποιο πρόβλημα εκεί. Όχι, κανένα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να σταματήσουμε επιτέλους να ε, ε, ε, λειτουργούμε σε βάρος των παρόντων. Να ψηφίσουμε τώρα, να μην περιμένουμε 10 λεπτάκια επειδή κάποιος λείπει. Πολύ ωραία. Ε, ε, το ψηφίζουμε λοιπόν και εγκρίνεται ομοφόνος. Ψηφίζουμε ε, σε μπλοκ τις 98 τροπολογίες που υπέβαλε η ΚΟΕ. Άρα πρέπει να είναι επίσημη η ψηφοφορία, να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες της ψηφοφορίας σας. Ε, την έναρξη της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τις 98 τροπολογίες. Υπέρ. Είναι αυτοί που δηλώνουν θετική ψήφο και όσοι είναι κατά δηλώνουν αρνητική ψήφο. Μπορείτε επίσης και να απέχετε. Πέρα της ψηφοφορίας. 18-2 και τρεις αποχές. Απορρίπτονται οι τροπολογίε αυτές. Επομένως, για το ψήφισμα. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Την 1. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ποιος ε, απέχει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. 17 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Πάμε τώρα στο θέμα της κινητοποίησης ε, του εργαλείου ευελιξίας. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια. Όχι, υπάρχουν δύο αποχές, συγγνώμη. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις προκαταβολές για το 2019. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ. Καμία κατά μία αποχή για το Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και για το Ταμείο Συνοχής. Προφορική τροπολογία για την τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται 24. 25. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. 4 και 3 αποτελούν αντικείμενο μίας ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Άποχες θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 16 ψηφί υπέρ, 7 κατά, 1 αποχή. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 και 5. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 17 ψήφοι κατά, 8 υπέρ. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Όχι, τροπολογία 21, ζητώ συγγνώμη. «21 υπέρ κατά». Η συμβαστική 1 υιοθετήθηκε. Η 21 άρα καταπίπτει. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Καταπέ... Καταπίπτει γιατί οθετήθηκε 21. Για το πρώτο μέρος της 21. Ποιο, ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους της τροπολογίας 21. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 θα το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51, 54 και 22. Τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 56. Υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 25 υπέρ μία ψήφος κατά μία αποχή συγχαρητήρια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 Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, μία κατά δύο εποχές. Συγχαρητήρια στο Γιάννη Γκάγερ. Πρόταση για τη ρύθμιση των συνόρων με ακτοφυλακή και σύνοριοφυλακή. Έκθεση Γιάννης Γκάγερ. Τροπολογίες 1, 2 και 3. Τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασα. 15 υπέρ, 12 κατά, χωρίς αποχές. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 για τα παραρτήματα υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την, ψηφο... την τροπολογία 15 για τα παραρτήματα. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 κατά, 11 υπέρ, μία εποχή. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 7 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει. Και η 11 το ίδιο. Η 8, τροπολογία 8, υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. 21 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή συγχαρητηρία στον εισηγητή. Για τις κοινέ διατάξεις. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για μια σειρά ταμείων και για την έκθεση Μούρεσαν. Δεν έχουν υπάρξει συμβαστικές τροπολογίες, αλλά ψηφοφορίες σε μπλοκ, ομαδικές, για να είμαστε συνεπείς στη δράση μιας. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, να θεωρήσω ότι υπάρχει συμφωνία να ψηφίσουμε με αυτόν τον τρόπο για να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των ε, ψηφισμένων κειμένων. Έχουμε λοιπόν τροπολογίες 27, 38, 40, 41, 62, 125, 192, 31, 36 κλπ. όπως βλέπετε. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα, τροπολογία 43, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε όνομα. Ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ 9 κατά. Ή 45. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 21 κατά 5 υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι για να σας βλέπω. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουν σηκωθεί όλα τα χέρια. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Έχουμε ένα δεύτερο σύνολο που καλύπτει τις 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 και 63. Γι' αυτό το σύνολο ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπθηκε. τροπολογία 62 που μπορεί να ψηφιστεί γιατί 63 απερίφθη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 και 69 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά δεν είναι προφανές οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 71 πέρας απορρίπτεται 15 ψήφοι κατά. Έναντι 13. 72 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 ε, υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 κατά πίπτη, 76 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται αλλά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 76. Τέλος, εγκρίνεται. 16 ψήφι υπέρ, 12 κατά. 77 καταπίπτει. 78 και 79, 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 κατά πίπτη 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας απορρίφθηκε 87 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 87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 94 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 94 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ, ενάντια 13 κατά. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99. Πέρασε. Εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ έναντι 9. Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά τροπολογιών 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Unblock υπέρ κατά αποχές καταπίπτουν. 107 υπέρ κατά. Δεν κατάλαβα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 107. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ έναντι 10 κατά. Σειρά τροπολογιών 108 μέχρι 113 unblock. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 116 είναι συμβατή με την 114 116 λοιπόν υπέρ κατά αποχές ε, ε, απορρίπτεται 117 κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 μέχρι και 132 unblock υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 μέχρι και 147 μπλοκ υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώθηκαν όλα τα χέρια άρα λοιπόν θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 148 άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται 17 ψήφι υπέρ. 149 υπέρ. Κατά. Δεν, καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπω να σηκώνονται πολλά χέρια. Λοιπόν, 149 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Εγκρίνεται. 19 ψήφι υπέρ. 150 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές δεν καταλαβαίνω γιατί πάλι δεν σηκώνται όλα τα χέρια ηλεκτρονικός έλεγχος για την 160 άρχεται τέλος απορρίπτεται αλλά παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας γιατί έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη την ώρα ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 5 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι 166 και οι 7 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 και 8 από κοινού ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά, ε, υπέρ αποχές απορρίπτεται, 175, 178 με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 37 έχει καταπέσει, η 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά δεν καταλαβαίνω καλά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 182. Τέλος. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία βλέπετε τι γίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Α, έχει καταπέσει. 185 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές κρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στα εκτιμώντας 28 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ έναντι 14 κατά για την 28 ήταν αυτό και τώρα έχουμε τη συμβιβαστική παριθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε για την 34 με ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ εναντί 3 κατά με δύο αποχές συγχαρητήρια στην κύριο Μορεσάν. Alors, nous en venons maintenant à l'instrument de coopération. Περνάμε τώρα στο μέσο εξωτερικής συνεργασίας. Έκθεση Καρδιά Ζαπάλ, Ρουμπιάλ, 11 υπέρ κατά αποχές 89 ε, ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογίες 12, 13 μέχρι και 23 unblock. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα έχουμε μία σειρά τροπολογίες που καταπίπτουν οι 90 μέχρι και 90 91, 92, 33, 95, 97, 98. Σύμβαστική α υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική α. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 94 ψήφοι έναντι... 14 με συγχωρείτε, έναντι 12 κατά. Τροπολογίες 25 και 65 από κενό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 26 υπέρ κατά επαληθεύμα με ηλεκτρονικό έλεγχο για την 26. Πέρας. Καταπίπτει. Ισοψηφία. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ Κατά. Επαληθεύουμε για την 30. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 29 υπέρ κατά Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, 32 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται, 33 και 66 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 35 υπέρ κατά αποχές Παληθεύουμε ηλεκτρονικά την 35. Απορρίφθηκε. 13 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Η 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά έχουμε τις τροπολογίες 67, 68, 69, από κοινού ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε με ηλεκτρονικό έλεγχο. Σκουτάν et ε, κλού. Τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά α, έχει καταπέσει 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 38 Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 14 υπέρ. 12 κατά. Το 38. 101. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε την 101. Πέρας. Απορρίπτεται 15 κατά 12 υπέρ. 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού ψηφίζουμε την 41. Πέρασα. Πέρασε, λέμε. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές θα το ψηφίσουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13-13. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 106. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά για τη 45. Ποιος είναι υπέρ της 45. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά ψηφίζουμε την 109 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 48 πέρασε απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές το επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 111. Πέρασε. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113. απορρίπτεται. 51 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Συγγνώμη, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 και 55 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις 81 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 81. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώθηκαν όλα τα χέρια. Ψηφίζουμε την 1. Πέρας. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά το επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 82. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 4. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την 84 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Πιστεύετε ότι θα έχουμε την ίδια πλειοψηφία για όλα? Και άρα ότι απορρίπτονται όλες? Όχι απαραίτητα. Άρχεται η ψηφοφορία για το 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική β, ποιο είναι υπέρ. Γάμα μάλλον, το σε, συγγνώμη, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 80 με την προφορική τροπολογία που τη συνοδεύει. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 κατά 12 υπέρ. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ. Δύο κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στο Χάιντερ. Έχουμε τώρα αλλιευτική συμφωνία μεταξύ της ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για το σύνολο του κειμένου. Έχουμε μία πρώτη ψηφοφορία για τη συμφωνία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έχουμε και μία ψηφοφορία για την απουσία γνωμοδότησης. με ονομαστική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση της κυρίας Χαουτάλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Χάουταλα. Έχουμε τώρα μία έκθεση για την αλληλευτική συμφωνία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαρόκου, έκθεση Φερνάντες και τροπολογία της κυρίας Χαουτάλα. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας, ποιος είναι κατά, απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε επί της συμφωνίας, υπέρ, κατά, αποχές. Και τώρα για τη γνωμοδότηση <coughs> με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Φερνάντες. Για το τμήμα 3 δεν υπάρχουν αιτήματα μεταβίβασης. Για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Έχουμε τρία αιτήματα μεταφοράς και μεταβίβασης. Θέλετε να μας εξηγήσετε την ε, εκτίμησή σας. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις μεταφορές. Τέσσερι μεταφορέ. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Απλά θέλω να σα ενημερώσω. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρότεινε να μεταφέρουμε 681.000 ε, ε, ευρώ για τον αγορά του εξοπλισμού. Βρέθηκαν εξοικονομήσεις από τις, ε, από τις μισθοδοσίες και λόγω του ότι ο πληθωρισμό κινήθηκε σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα. Άρα η ε, ε, προσαρμογή των μισθών ήταν χαμηλότερη. Δεύτερη μεταφορά αφορά 9,7 εκατομμύρια ευρώ προς ε, την κατασκευή ενός τρίτου πύργου για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η εξοικονόμηση επίσης προήλθε από την μυθοδοσία για τους ίδιους λόγους όπως είπα και πριν, αν και βρέθηκαν και άλλες εξοικονομίες μέσω μισθώσεων leasing, αυτοκινήτων και άλλων ε, οδών. Η ΕΙΕΔ έχει ένα αίτημα για 12,5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν ένα νέο κτίριο στην ε, Ουάσιγκτον το οποίο θα αγοράσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και υπάρχουν κάποιες μικρότερες μεταφορές ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξοπλισμό ασφαλείας οι μεταφορές αυτές είναι χαμηλότερες. Υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, χαμηλότερος πληθωρισμός, από εκεί προέρχονται οι εξοικονομήσεις αυτές. Και τέλος, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποεκτίμησε τις κτηριακές του δαπάνες λόγω υψηλότερων εξόδων για, για εξοπλισμό ασφάλειας κτλ ε, όπως και για διερμηνία, μετάφραση, πληροφορικά συστήματα και εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτές οι μεταφορές ανέρχονται σε 200.000 ευρώ και επαναλαμβάνω ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για καμία από αυτές τις μεταφορές. Συστήνω να τις εγκρίνουμε. Ευχαριστώ κύριε Σίτα. Θέλουν οι σκιώδεις να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω κανείς να ζητά το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Δοσάντος. Ε, ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, μόνο για να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο εισηγητής, ακόμα και αν δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένο με τα πληροφορίε που έλαβα όταν τις ζήτησες. Αλλά αυτό βεβαίως δεν αρκεί για να αντισταθώ ή να αντιτεθώ στα όσα ψηφίζουμε. Θα υπερψηφίσω την πρόταση. Merci. Σας ευχαριστώ. Θέλει άλλο το λόγο? Όχι. Ο εισηγητή μας ε, μας λέει ότι εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνονται αυτές οι τροπολογίες. Εγκρίνονται λοιπόν και τώρα το λόγο έχει η Μόνικα Χολμάιερ την οποία συγχαίρω για την επανεκλογή της, γιατί θα είναι γενική εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό το τμήμα 3 για τον προπολογισμό του 2020. Να συγχαρώ και τον κύριο Μάνκα που θα είναι εισηγητής για τα άλλα τμήματα. Έχετε το λόγο για τα κτίρια. Και συγκεκριμένα στην Πρετόρια για το πράγμα για το οποίο μας έχετε μιλήσει. Λοιπόν, για την αγορά του κτηρίου στην Πρετόρια, η μετακόμιση οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ούτε δυνατότητες επικοινωνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου οχημάτων, προσώπων, τα κουφώματα δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφαλείας και δεν υπάρχει δυνατότητα περίφραξης του κτηρίου. Ε, τα μέτρα ανακαίνησης ε, θα ήταν ε, πάρα πολύ δαπανηρά και το κτίριο δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή περιοχή της πόλης. Λάβαμε 21 προσφορές. Το νέο κτίριο χτίστηκε 2004-2005. Έχει 130 ε, μάλλον 300 ε, τετραγωνικά μέτρα έκτασης γραφείων. 24 από αυτά προβλέπονται να παραδοθούν στην ε, ΕΤΕΠ. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει το κόστος για την αγορά του ακινήτου ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ και πάρθηκε η απόφαση πέρα αυτού του κτηρίου. Να μην μακρηγορήσω, θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για το ποιος ακριβώς είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του κτηρίου, έχω τις πληροφορίες πλέον αυτές, μπορείτε να τις ε, έχετε, τις, ε, μπορώ να σας τις θέσω και στη διάθεσή σας αν τις επιθυμείτε. Εγώ προτείνω να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Voulez-vous nous présenter également le projet pour l'Azerbaïdjan? Oui. Θέλετε να μας παρουσιάσετε και τις ε, προτάσεις. Ναι, για το Αζερβαϊτζάν. Εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι ο ιδιοκτήτη ενό κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον 11ο όροφο, ενό κτηρίου στο οποίο στεγάζονται και η πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς και άλλες υπηρεσίες και διεθνεί οργανισμοί, ε, μισθώνεται για 81 χρόνια. Πληρώνουμε 5 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό και με αυτό το αντίτιμο, αντίτιμο θα έχουμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο κτίριο για 81 χρόνια. Από το 10ο χρόνο θα έχουμε αποσβέσει τα, τα, έξοδα, τα αυτά. Μου κάνει εντύπωση. Ε, είναι πάρα πολύ χαμηλό το, ε, ε ενίκιο που μας ζητά ο ιδιοκτήτης, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αφού είναι τόσο οικονομική η πρόταση αυτή που λάβαμε, ε, εμείς δεν έχουμε παρά να την αποδεχτούμε αυτή την πρόταση. Σε περίπτωση που μάλιστα ε, αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε το κτίριο πριν από την εκπνοή των 81 ετών, θα λάβουμε πίσω και το αντίστοιχο ενίκιο που δεν θα έχουμε ε, ε, αξιοποίηση των χρόνο, δηλαδή για τον οποίο δεν έχουμε ε, περάσει μέσα σε αυτό το κτίριο. Οπότε επειδή είναι μια καλή πρόταση θα πρότεινα να υπερψηφίσουμε και αυτήν. Ευχαριστώ. Άλλες παρατηρήσει Ποιος θέλει το λόγο. Ε, αν δεν θέλει κανείς το λόγο θα συνεχίσουμε με την ονομαστική ψηφοφορία για την Πρετόρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 12 υπέρ, 1 κατά. Δεύτερη ψηφοφορία για το Αζερβαϊτζάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι φάκελοι για τα κτηριακά. Δεν υπάρχουν άλλες επικοινωνίες, ανακοινώσεις. Όχι, συγγνώμη, παρακαλώ. Προσπαθούμε ακόμη να καταλάβουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κτηρίου ε, της ε, πρεσβείας μας στην ε, Μόσχα. Έχουμε ένα όνομα, όμως μεσολαβούν και τρεις εταιρείε. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώ ακόμη αν πράγματι το όνομα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κτηρίου. Ε, λέω λοιπόν να επιμείνουμε λίγο, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο σαν κούκλα μ, μπάμπουσκα. Ε, δεν θέλω να ξέρω μόνο ποιος ε, μπαίνει μπροστά, ποιος είναι στη βιτρίνα ε, αυτής της μίσθωσης. Θέλω να ξέρω σε ποιον πραγματικά θα καταλήξουν τα χρήματα. Mm, έτσι δεν είναι. Είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από την ε, ε, Κύπρο. Ε, υπάρχουν δύο δικηγορικά γραφεία, δύο εταιρείες και εκείνος που διαμένει, ε, το, το άτομο που γνωρίζουμε και υποτίθεται ότι διαμένει στην Κύπρο, αλλά δεν έχουμε λάβει νόμιμα έγγραφα που να πιστοποιούν κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την, ε, με επιμονή να δούμε ποιο ακριβώς θα μάθουμε. Γιατί εμφανίζεται διαρκώς ένα συγκεκριμένο όνομα, αλλά μόνο ως διευθυντής των εταιριών που εκπροσωπεί που εκπροσωπούν τον ε, ιδιοκτήτη. Ε, δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι ο πραγματικό οικονομικό δικαιούχο και ποιο είναι ο κάτοχο αυτού του κτηρίου. Ε, ε, θα υποστηρίξω λοιπόν με αποφασιστικότητα το αίτημά σας, διότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωκοινοβουλίου να καταστεί ύποπτη για συνενοχή σε φορολογικές ε, βελτιστοποίησεις. Είμαστε κατά. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εμπλακεί η Ευρώπη σε τέτοιου είδους ε, ε, διαδικασίες. Και ξέρω πως κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πρότυπο ακεραιότητας και σεβασμού των κανόνων της διαφάνειας. Ο κύριος Γιούνκερ τα είπε αυτά. Πολύ ωραία. Εάν δεν έχετε ερωτήσεις υπό τα διάφορα, θεωρώ ότι... Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και την ημερήσια μας διάταξη και να διευκρινίσω μόνο ότι προγραμματίσαμε την 5η το πρωί στις 13 Δεκεμβρίου κοινή συνεδρίαση Badge Cont για τις επενδύσεις στο κράτος δικαίου και Μπούτζ Έκον για το InvestEU. Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών, θα συνεδριάσει του χρόνου στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Pas δεν θα κάνουμε άλλε συνεδριάσει λοιπόν τη Επιτροπής προπολογισμών από ότι αυτές τις κοινέ και επειδή έχω θα λείπω την Πέμπτη το πρωί θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και να σας πω πως ε, πολύ αξίζετε αυτή την ε, χειμερινή, το χειμερινό διάλειμμα. La séance est levée. Πέρα συνεδρίαση.